μέχρι τις 12 το βράδυ. Ε, δεν μου απομένει παρά να ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους ε, λίγη αλλά ιδιαίτερα προσεκτική. ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και λίγη η τελευταία μου προεδρία νυχτερινής συνεδρίασης. Ε, ε λίγη λοιπόν η συνεδρίαση για σήμερα.